εστίασης έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Α, για διαδικαστικό ο κύριος Λιμπέρο Κάστρο ε, ζητάει το λόγο. Σας ακούω κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους.